των υποθέσεων θα επαληθεύσει τα, τις αρμοδιότητες του κυρίου Ζάμε Ντίμετς, του κυρίου Μάθιους, του κυρίου Ζαμέ και του κυρίου Ράτκε και Μπούλοκ για να επικυρώσει τις ε, εντολές που έχουν λάβει από τις... Ε, και ε, επικύρωσε μάλλον, συγγνώμη, την εντολή που έλαβαν στις 24 και 29 Ιουνίου